ερήσια διάταξη να περάσουμε στο δεύτερο θέμα ε, για την πολιτική συνοχή μετά το 2013. Θα δώσω το λόγο καταρχήν ε, στη συντάκτρια, την κυρία Ντανούτα Μαρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Πίτροπη, ε, συνάδελφοι. Πριν από τρία χρόνια εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική λαμβάνοντας υπόψη την ε, μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βέβαια πρόκειται για μια σοβαρή πρόκληση και η πολιτική συνοχής προέβλεπε τις κλιματολογικές αλλαγές στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνες, αποτελεσματικότητα σε διάφορους ε, τομείς και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ε, πολιτική συνοχής ε, θα μπορούσε να περιέχει όλα τα θέματα που υπάρχουν τώρα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 διότι ο στόχος μας είναι να προκαταλαμβάνουμε την αλλαγή και όχι να την ακολουθήσουμε και γι' αυτό είχαμε δημοσιεύσει ένα αναλυτικό αναλυτικό, ε, μια αναλυτική έκθεση και τώρα είμαστε έτοιμοι για να ε, επιλύσουμε τα προβλήματα του μέλλοντος. Έχουμε διαθέσει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ιδίως στην, ε, το συνδυασμό μέσων για την επίλυση της οικονομικής κρίσεως και για την αλλαγή του περιβάλλοντος. Αλλά το βασικό είναι το μέλλον, κύριε Πρόεδρε, διότι στο θα χρειαστούμε μία ισχυρή συλλογική αντιμετώπιση από τους πολίτες οι οποίοι τώρα είναι πληροφορημένοι, γνωρίζουν πολύ καλά τι διακυδεύεται όταν λαμβάνουν τη μία ή την άλλη επιλογή και αυτό το βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις. Ο Ζακ Ντολόρ είχε πει κάποτε ότι η ενιαία αγορά αναφέρεται στον ανταγωνισμό, ότι ενισχύει την αποτελεσματικότητα και ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει η ενιαία αγορά να λειτουργήσει και η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να βασιστεί ακριβώς σε αυτές ε, τις ε, δυνατότητες θα πρέπει να ε, κινητοποιήσουμε όλες τις περιφέρειες και τις περιοχές διότι η πείρα μας μας απέδειξε ότι η κινητοποίηση αυτή είναι πλέον αποτελεσματική ε, αν ε, υπάρχουν, υπάρχει εφαρμογή του κώδικα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Έχουμε ήδη περάσει τη δοκιμασία της επικουρικότητας που λειτουργεί για την Ευρώπη. Η μεταρρύθμιση του 2006 για την πολιτική συνοχή επιτρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ της ε, προσθετικότητας ε, και ε, της χρηστής διακυβέρνησης και πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις προσπάθειες διότι η επικουρικότητα ήδη ήδη βασίζεται στην πολιτική και αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, ιδίως στο τοπικό επίπεδο, διότι όσοι θεωρούν ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να περιοριστεί στις Βρυξέλλες ή στις πρωτεύουσες ή δεν καταλαβαίνουν ή δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, διότι η Ευρώπη επιζητεί κοινού στόχους και ε, ε, δεν είναι σωστό να αποφασίζει για όλα τα οικονομικά θέματα. Η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να μας διαιρεί, θα πρέπει να είναι μια πολιτική για όλους. Και εφόσον ε, η, εσωτερική αγορά ιδίω ε, ε, είναι αυτή η οποία είναι. Και το ενιαίο νόμισμα μας βοηθά στην αλληλεξάρτηση, είναι κοινό ευρωπαϊκό Έχουμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε αποτελέσματα και θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με το κοινό. Ε, χρειάζεται μία πολιτική ανάπτυξη, χρειάζεται μία πολιτική συνοχή η οποία να είναι ε, εξελικτική και στην οποία να εμπλέκονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή η Ευρώπη χρειάζεται νέα ενέργεια για να μπορέσει να ανανεωθεί και να ανανεωθεί επικοδομητικά. Το ερώτημα είναι από πού πρέπει να προέλθει αυτή η ενέργεια, διότι για μένα αυτό σήμερα είναι σαφές. Η ενέργεια πρέπει να έρθει από τα κάτω. Θα πρέπει δηλαδή να οφείλεται στην άμεση εμπλοκή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης προς όφελος των, ε, της επιτεύξεως των ευρωπαϊκών στόχων. Σας ευχαριστώ. Τώρα, εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει ο κύριος Δαμέσκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτές, οι ερωτήσεις ήταν πολύ εύστοχες και υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχή, καθώς επίσης και την αφοσίωση που έχετε στο θέμα αυτό ε, σαν μέρος της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αναφερθήκατε στην ε, διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων που έχει αναγνωριστεί σαν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς. Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση στην Ευρώπη τονίστηκε από το έγγραφο διαβούλευση ε, που παρουσίασε η Κομισιόν για τη στρατηγική για το 2020. Η πολιτική συνοχή είναι ένα καλό παράδειγμα ε, διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων. Είναι ένα σύστημα διακυβέρνηση που αξιοποιεί τι τοπικέ και περιφερειακέ γνώσει σε συνδυασμό με τι στρατηγικέ κατευθύνσει που δίνονται σε κοινοτικό επίπεδο και συντονίζει τι παρεμβάσει ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση. Τα ισχυρά σημεία τη διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων επίση ε, τονίστηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών στο Λευκό Βιβλίο του Ιουνίου του 2009, όπου καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τα διάφορα επίπεδα τη ε, διακυβέρνηση και ε, να εφαρμόσει μια πολιτική συνοχή που θα συμβάλλει στην επιτυχία και των άλλων πολιτικών. Για τα δύο θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη εγκατάλειψη του στόχου 2 και την επιλεξιμότητα όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών, Κατά την περίοδο 2007-2013 όλες οι περιφέρειες είναι επιλέξιμες για υποστήριξη από, τα περιφερειακά, από το Περιφερειακό Ταμείο. Μετά από το 2013 δεν υπάρχει επίσημη θέση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την τρίτη σας ερώτηση για την αποδυνάμωση της αρχής της προσθετικότητας. Η προσθετικότητα είναι μία από τις βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής. Εξασφαλίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δεν υποκαθιστούν ε, δημόσιες ή άλλες ισοδύναμες δαπάνες των κρατών μελών. Έτσι εξασφαλίζεται ε, μία πραγματική ε, ε, επιρροή των παρεμβάσεων των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής συνοχής μετά το 2013, η συνθήκη της Λισαβόνας διατηρεί το στόχο της μείωσης των ανισοτήτων ε, στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη μάλλον των διαφόρων περιφερειών και την υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών στο άρθρο 174. Επιπλέον, το άρθρο 176 επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη έχει σκοπό να βοηθήσει να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες οι περιφερειακές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ε, προσαρμογών των περιφερειών που παρουσιάζουν ε, υστέρηση και μέσω της ε, σύγκληση των ε, βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή. Όσον αφορά τώρα την πολιτική συνοχή μετά το 2013 και την επόμενη ερώτηση, θα ήθελα ε, και πάλι να επιστήσω την προσοχή σας στο έγγραφο διαβούλευση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 που επιζητά ε, ενεργό υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων όπως είναι η κοινωνική εταίρη και η κοινωνία των πολιτών και αναγνωρίζει ότι το όραμα του 2020 για να περάσει ε, πρέπει να περάσει σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε επιτυχία η Κομισιόν δεν έχει ακόμα αναπτύξει τη θέση σχετικά με το ρόλο τη πολιτική συνοχή στη στρατηγική για το 2020. Όμω η πολιτική συνοχή έχει την ικανότητα να κινητοποιήσει τοπικού και περιφερειακού ε, παράγοντε ε, για την επιδίωξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για την ερώτηση σας αν η Κομισιόν έχει σκοπό να δημοσιεύσει μια λευκή βίβλο για την πολιτική συνοχή. Δεν προβλέπεται για την εδαφική συνοχή ε, κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχει όμως, υπάρχουν τα συμπεράσματα της πράσινης βίβλου για την εδαφική ε, διάσταση που θα περιληφθούν στην ανακοίνωση για μετά το 2013 και την ε, πέμπτη έκθεση και που θα υποβληθούν το 2010. Για την ερώτηση σχετικά με το ρόλο ε, του Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην πολιτική συνοχή, η απάντηση είναι ότι η πολιτική συνοχή διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο για την πραγματοποίηση των ε, ε, προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που θα συνεχίσει να επιδιώκει του στόχου του σύμφωνα με τον τίτλο 11 τη Νέα Συνθήκη. Η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή ε, απαιτεί ένα μείγμα πολιτικών σε διάφορα επίπεδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι πολιτικές του είναι ε, μια σημαντική διάσταση όλων αυτών των ε, προσπαθειών. Όσον αφορά το ρόλο της πολιτικής συνοχής σε σχέση με τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική συνοχή προσφέρει πραγματικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Η Κομισιόν σε μια ανακοίνωσή της του 2008 υπογραμμίζει πόσο σημασία έχει η πολιτική συνοχή για την ε, πραγματοποίηση των στόχων της Λισαβόνας, επενδύσεις, ε, ε, υποδομές κλπ. Η Κομισιόν εστιάζει στο γεγονός ότι η εφαρμογή του σχεδίου επενδύσεων μπορεί να συμβάλλει και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία ανάμεσα στι ε, υπηρεσίε τη Κομισιόν και τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Ένα πρακτικό παράδειγμα ε, συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τη Κομισιόν είναι ο οδηγό που δημοσιεύθηκε το 2007 για τι επενδύσει και ε, στην καινοτομία όπου παρουσιάζονται όλες οι δυνατότητες που δίνουν τα τρία ε, ταμεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά δε ε, την σύνδεση ανάμεσα στις ε, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οικονομική υποστήριξη. Αυτό εξασφαλίζεται και από το Συνισμό της, πολιτικής συνοχής και της ε, πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου, όπως ε, το υπογραμμίζουν εξάλλου οι κατευθυντήριες γραμμές και για τα δύο αυτά είδη πολιτικής. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας και ε, περιμένω να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι πολιτικές ομάδες. Θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Βανίστερόη. Ο κύριος Νίστερ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρόκειται εδώ καταρχήν για την επί της ουσίας αξιολόγηση και της πρόοδου της πολιτικής σύνοχης. Θέλουμε φυσικά και στην ενδιάμεση αναθεώρηση ως κοινοβουλίου να ε, εμπλακούμε και να δούμε τι θα γίνει με την πολιτική συνοχή μέχρι το 2020. Είναι ένα κέριο θέμα αυτό. Προς μεγάλη μας έκπληξη έπρεπε να διαπιστώσουμε όμως ότι από πλευράς ε, αξιολόγησης επί της ουσίας στο non-paper για την προπαρασκευή της ενδιάμεσης αναθεώρησης δεν γινόταν καθόλου λόγος ε, γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν η νέα Επιτροπή ε, την επί της ουσίας αποτίμηση πρέπει να την υποβάλει. Δεν είναι αποδεκτό ότι έτσι απλά και μόνο μια επιφανειακή παρουσίαση, σταχυολόγηση γίνεται εδώ για την πολιτική συνοχή. Θέλουμε περισσότερη ανάπτυξη, θέλουμε την πράσινη ανάπτυξη και την ε, προώθησή της. Αυτό το είχε προναγγείλει ο Μπαρόζο. Θέλουμε μια περιφερειακή πολιτική στην Ευρώπη που θα λειτουργεί ε, ενοποιητικά και μέσα σε ένα πλαίσιο ολοκλήρωση. Ε, οι συνθήκε τη Λισαβόνα, οι κλιματικέ αλλαγέ, ε, πολλά γίνονται στι περιφέρειε και πρέπει να υποστηρίξουμε αυτέ τι περιφερειακέ πρωτοβουλίε. Πρόκειται για τα σημεία πυρήνε και την ίδια την καρδιά τη στρατηγική μα. Πρόκειται για όλε τι περιφέρειε λοιπόν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και κάποια γενικόλογη αναφορά στην Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βλέπουμε ότι στις πλούσιες γίνεται, προωθούνται οι πλουσιότερες περιφέρειες. Αυτό δεν πρέπει να ε, επιτρέπεται. Πρέπει τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι λανθασμένο να βοηθάμε μόνο ε, κάποιους και όχι εκείνους που χρειάζονται τη βοήθεια. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης ε, είναι τεράστια σημασία στα περιφερειακά κονδύλια. Δαπανώνται γρήγορα και χρησιμοποιούνται άμεσα. Το 2009 στην Νότια Ολλανδία, για παράδειγμα, στην δική μου ε, περιοχή, πάνω από ε, ε, μπορούμε να πούμε ότι 100% για την καινοτομία και τους νέους στόχους χρειάζονται τα κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν για τα περιφερειακά κονδύλια να δούμε τη σωστή τους χρήση. Και μια άλλη ερώτηση προς τον Επίτροπο. Είπατε σε σχέση με την ε, περιφερειακή συνοχή. Εδώ όμω εμείς ως ε, Κοινοβούλιο έχουμε συναπόφαση, δικαιώματα συναπόφασης και αναμένουμε να ληφθεί υπόψη αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέλ παρακαλώ θα ε, παρέμβει στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ανέμενα μια πιο ενδιαφέρουσα εισαγωγή σε αυτό το θέμα διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή πραγματικά πρέπει να αλλάξει μετά το 2013. Έχουμε τελείως διαφορετικές προκλήσεις σήμερα πια σε σχέση με πριν από 10 χρόνια και για τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται στο προσκήνιο η αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε όλες οι περιφέρειες θα πρέπει στην πολιτική συνοχή να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει οποιαδήποτε προσπάθεια να επανεθνικοποιηθεί η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ε, καταδικαστεί και να καταγγέλλεται από πλευρά μας. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τους πολίτες αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια προσέγγιση που θα μπορούν οι πολίτες να ταυτίζονται με αυτήν. Για μας είναι αδιαμφισβήτητο ότι φυσικά πρέπει και εμείς να αλλάξουμε και να αλλάξουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Πολιτική συνοχή. Ποιες προτεραιότητες πρέπει να προαχθούν. Δεν είναι δυνατόν όλα, τα πάντα να προάγονται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρέπει να επιλέξουμε και να επικεντρωθούμε σε μια σωστή επιλογή για τις υποδομές, ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως τις κλιματικές αλλαγές, όπως τις δημογραφικές αλλαγές και θα πρέπει στο μέλλον να είμαστε πιο υπεύθυνοι με, τα, με την πολιτική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Πρέπει να είναι ένα έργο λοιπόν αυτό, ένα στόχος να επικεντρωνόμαστε όχι επειδή, στα αστικά κέντρα, όχι επειδή δεν θέλουμε να προσέξουμε τις περιοχές της Υπέτρου, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι 80% των πολιτών μας ζουν στις πόλεις και στον αστικό περίγυρο των πόλεων και ότι η ανάπτυξη των πόλεων δυστυχώς διαχωρίστηκε από την πολιτική συνοχή όσον αφορά τον, και τον τομέα της ε, πολιτικής γεωργίας για παράδειγμα. Εδώ να υπάρξει μια σωστή διασύνδεση και μια δικτύωση είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να θέσουμε αυτό το αίτημα, να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Τέλος, και για την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος νομίζω ότι δεν επαρκεί απόλυτα. Πρέπει να δούμε και την υποστήριξη των ίδιων των ανθρώπων που πρέπει να στηρίξουμε στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Τι σημαίνει αυτό για μας σε πρώτη γραμμή κυρίως κατάρτιση, εκπαίδευση, παιδεία, επιμόρφωση, επαγγελματικά προσόντα από την παιδική ηλικία μέχρι την ε, ηλικία που οι άνθρωποι πια συνταξιοδοτούνται και είναι ε, και υπερήλικες. Πρέπει να συνεχίσουν να επιμορφώνονται και να καταρτίζονται. Στον τομέα της πολιτικής συνοχής πρέπει αυτό να ενταχθεί και να μην παρεκκλίνουμε όσον αφορά για παράδειγμα την αποσύνδεση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής. Η διασυνοριακή διαμεθοριακή συνεργασία είναι σημαντική για μας. Θέλουμε να ενισχυθεί και αυτή και θέλουμε να απλουστευτούν οι γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέλ. Για τους Δημοκράτες Φιλελεύθερους για δύο λεπτά η κυρία Γιους Μινόβα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η συζήτηση για τα διαθωτικά ταμεία και τη μεταρρύθμιση τους έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει ικανά δημοσιονομικά μέσα, χρηματοοικονομικά μέσα που θα ανταποκρίνονται στο ανθρώπινο δυναμικό και τις ανάγκες του. Πρέπει να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε μια πολιτική συνοχή που θα διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών. Αυτή η πολιτική ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα μετρήσιμο και αξιόλογο στοιχείο για την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όμως υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές μεταξύ των επιμέρους ε, ευρωπαϊκών περιφερειών και υπάρχει και η τάση για περαιτέρω όξυνση αυτών των διαφορών. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιες περιοχές ίσως να απομονωθούν. Εκπροσωπώντας μία από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνω ιδιαίτερη έκκληση στο να προσέξουμε ιδιαίτερα τις περιφέρειες και περιοχές χαμηλού εισοδήματος Ταυτόχρονα κατανοώ απόλυτα ότι τα διαθροτικά ταμεία δεν είναι εκείνα τα οποία εδώ θα επαρκέσουν αποκλειστικά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους εσωτερικούς μας πόρους. Αλλά αν υπάρχει μια σωστή προσέγγιση από πλευράς μέσων και εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των στόχων, τότε αν δεν λάβουμε τα σωστά μέτρα θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει εδώ να δοθεί σε σχέση με χώρες που δεν, δίνουν, δεν ε, σημειώνουν επαρκή πρόοδο θα πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση της οποίας πρέπει να τύχουν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα διασυνοριακής σημασία. Έτσι οι χώρες που έχουν υψηλότερο και χαμηλότερο ΑΕΠ θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και τέλος η απασχόληση είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το πώς η πολιτική συνοχή συναρτάται με άλλες πολιτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομάδα των Πρασίνων και την Ελεύθερη Πράσινη Συμμαχία θα λάβει τον λόγο η κυρία Σρέτερ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μάλιστα κύριε Επίτροπε για το ποια σημασία τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή στην Ευρώπη είναι η ίδια η καρδιά, ο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτή είναι η πολιτική που η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρατά ενωμένη και είναι ένα σύμβολο αλληλεγγύης και ένα σύμβολο υπέρβασης ε, εθνικών εγωισμών. Είναι ένα μέσο και εργαλείο για όλες τις περιφέρειες. Και γι' αυτό εδώ Ευρωπαϊ... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης θα εγκαταλειφθεί ίσως. Γιατί αυτό δεν είναι υπέρ της χρηστής διαχείρισης. Όταν κρυφά, παραβίστο ε, παρουσιάζει, έχει κάποια στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσον αφορά τον μηχανισμό αλληλεγγύης για το πώς ε, όταν εμείς ζητούμε να συνεχιστεί η λειτουργία του δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που έχουμε παράδειγμα τις ε, αλλαγές του κλίματος, τις δημογραφικές αλλαγές ε, και όλα αυτά και βλέπουμε ότι έχουμε και δημοσιονομικά οικονομικά προβλήματα χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση αλλά μια μεταρρύθμιση πρέπει να είναι διαφορετική από αυτήν πρέπει να πετύχει μια υφορία στην ανάπτυξη στις περιφέρειές μας πρέπει τις περιφέρειές μας να τις στηρίζει για την υλοποίηση των προγραμμάτων και σχεδίων τους και όχι να ακολουθείτε μια προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω. Πρέπει σε πολύ στενή εταιρική σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους σε όλες τις περιφέρειες να υπάρχει μια συνέργεια. Γνωρίζουμε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε και τη μέθοδο για την προσέγγιση ε, κατά την ανάπτυξη της υπαίθρου μια εξαιρετική προσέγγιση με πολύ θετικά αποτελέσματα στην οποία προσέγγιση εμπλεκόντουσαν όλοι και πετύχαμε, πετυχαίναμε μεγάλη αποδοχή ε, στις περιφέρειες. Χρειαζόμαστε όμως γενναιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει ναι υπέρ του μηχανισμού αλληλεγγύης ώστε να καθορίζουν οι περιφέρειες τι είδους ανάπτυξη επιθυμούν και όχι αυτό να επιβάλλεται από τις εθνικές κυβερνήσεις μόνο και αποκλειστικά. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σρότερ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές για δύο λεπτά. Θα λάβει τον λόγο παρακαλώ Βλάσακ. Ευχαριστώ θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι η σημερινή πολιτική σύνοχης είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ακριβώς όπως μεταβάλλεται και η Ευρώπη μεταβάλλονται και τα κράτη-μέλη αλλάζουν και οι συνθήκες και όροι για αυτή την πολιτική το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 θέτει περισσότερα ερωτήματα από ότι δίνονται κάποιες απαντήσεις και αυτό αφορά την προώθηση και προαγωγή των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές, τεχνικές υποδομές ε, κτλ. Πρέπει επίσης η ποιότητα ζωής και διαβίωσης των πολιτών να βελτιωθεί. Πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Πρέπει επίσης ε, η διοικητική επιβάρυνση να μειωθεί. Είναι πράγματα στα οποία χρειαζόμαστε κατεπηγόντως απαντήσεις. Και για την μελλοντική ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλη σημασία. η πόλεις και τα αστικά κέντρα να διαδραματίζουν ρόλο στη διαχείριση των κονδυλίων και τα κονδύλια αυτά να στρέφονται στη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Σε αυτούς λοιπόν τους δύο τομείς θα πρέπει οι smart cities να προαθούν, οι πόλεις οι οποίες, ε, τις οποίες θα διαχειριζόμαστε με ευφυή τρόπο και θα ε, έχουν μια ευφυή προσέγγιση και στη δομή τους αλλά και στη διαχείρισή τους ώστε σύγχρονα συστήματα και ευφυής τεχνολογία και τεχνογνωσία να χρησιμοποιείται. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σε αυτό το τομέα στρατηγικές επενδύσεις είναι αναγκαίες και αυτό όχι μόνο στο επίπεδο των πόλεων και των αστικών κέντρων αλλά και στο επίπεδο των κρατών μελών και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Ένα ευφυές σύστημα ε, συγκοινωνιών ώστε να μην υπάρχουν συμφορήσεις και προβλήματα οχήματα και στενοποιεί στην κυκλοφορία. Να μπορεί κανείς να μετακινείται εύκολα. Αυτά τα συστήματα είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία και για τους πρεσβύτες πολίτες, τους ηλικιωμένους, να μπορούν και αυτοί να μετακινούνται με τον πιο καλό τρόπο η οικονομική κρίση ε, επισκιάζει τις συζητήσεις μας ε, και καθιστούν αυτά τα θέματα ακόμα περισσότερο σημαντικά από ό,τι σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να σκεφτούμε χρησιμοποιώντας τα κονδύλια που θα διατεθούν. Σας ευχαριστώ για την Ενωτική Αριστερά. Θα λάβει τώρα τον λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η πολιτική συνοχή της ευρωπαϊκής ένωσης όχι μόνο δεν έχει μειώσει περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες αλλά έχει συμβάλει στην όξυνσή τους. οι τιμές που δίνουν οι στατιστικές είναι πολλές φορές πλασματικές κάτι που και η ίδια η ευρωπαϊκή ένωση αποδέχεται γι' αυτό και δημιούργησε το καθεστώς μεταβατικής στήριξης για σειρά περιφερειών τρεις από τις οποίες βρίσκονται στη χώρα μου στην ελλάδα. ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης στο καπιταλιστικό σύστημα είναι αδυσόπιτος ιδίως σε περιόδους κρίσης που οι αντιθέσεις οξύνονται ακόμα περισσότερο και δυστυχώ οι προβλέψει για το 2013 είναι ακόμα πιο δύσκολε για του εργαζόμενου, ιδιαίτερα στι λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ. Η πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει να εξοραίσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, να εξαγοράσει συνειδήσει, να αποπροσανατολίσει του εργαζόμενου και κυρίω να εξασφαλίσει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η επιδίωξη προσωρινή εξισορρόπηση αντιθέσεων μεταξύ τμήματων τη πλουτοκρατία που ονομαζόταν κύβδηλα αλληλεγγύη αντικαθίσταται πλέον από τον κανόνα του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και στην στρατηγική της λισαβόνας και στην στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης για το είκοσι Αυτό απαιτεί νέε μορφέ περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση, όπω προτείνουν στην Ελλάδα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, διευρυμένη ε, αμεσότερη παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα περιφερειακά όργανα, διαφορετική εδαφική συνεργασία που θα υπερβαίνει και αυτά τα εθνικά σύνορα. Εμεί καλούμε του εργαζόμενου να απορρίψουν αυτή την πολιτική και αξιοποιώντα αυτή την παρέμβασή μου θα ήθελα να σα παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε να ασκήσετε το βάρο σα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οι οποίοι βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγγουράκη. Για τέσσερα λεπτά τώρα στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μπάφτον παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Όσο αναφορά την πολιτική συνοχή ε, και την, ε, και την πρόταση προβλέπεται ότι θα αλλάξει η κατανομή και ε, ο έλεγχος σε τοπικό επίπεδο θα είναι αντίθετος εις ε, τις ε, αρχές διακυβέρνησης για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι κοινέ διαρθρώσεις. Η επιστροφή στα κράτη-μέλη θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ε, κατανέμουν εθνικά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη ε, ε, που είναι νέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν χαμηλή, χαμηλές απολαβές, πράγμα το οποίο θα διτηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να χρηματοδοτεί μαζί με άλλα πλούσια κράτη όλο και περισσότερο τις ε, αδύναμες χώρες. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τόσοι υποψήφοι να προσχωρήσουν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να δίνετε τέτοια βοήθεια στα νέα κράτη διότι η ε, Νορβηγία και η Ελβετία δεν πλησιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνουμε και να μην παίρνουμε τίποτα ε, πίσω. Ε, θέλουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ομοσπονδία αλλά η πολιτική συνοχή στην οποία βασίζεται η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει απολαβές σε όλα τα μέλη της και σιγά σιγά εγκαταλείπεται η συνεργασία μέσω μιας παγιοποίησης πρέπει να υπάρχουν στενότερες σχέσεις στην αγροτική πολιτική υπάρχει όλο και μία μεγαλύτερη γραφειοκρατία στην Ευρώπη και ε, ε, αυτά είναι η βάρος της στρατηγικής και ορισμένων κρατών που ε, πληρώνουν περισσότερα από ό,τι παίρνουν όπως το Ενωμένο Βασίλειο. Έχουμε διάφορα προγράμματα και για τα οποία είχαμε ζητήσει ζητήσει πόρους και ε, εις ε, την Ουαλία παραδείγματος χάνει χρηματοδότηση θα δοθεί πολύ αργότερα και δεν ε, υπάρχει καμία πληροφόρηση για το πότε πρόκειται να χρηματοδοτηθούν τα τοπικά μας προγράμματα πράγμα το οποίο θα αποξενώσει ακόμη περισσότερο τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στην άνοιξη στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλό θα ήταν να γνωρίσουμε τι γίνεται σε όλα τα κράτη-μέρη και οι επιπτώσεις εις την Ουαλία σημαίνει ότι θα επηρεάσουν την κατάσταση στην περιοχή μας και τα προγράμματα που καταρτίζονται και αν είναι να έχουν ευεργετικό και επίπτωση στην περιοχή μου υπάρχει αρνητική. Η μείωση της χρηματοδότησης στην Ουαλία θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα και τον γεωργικό τομέα. Άρα τώρα είναι η στιγμή κύριε Πρόεδρε να υπάρξει μια δημοσκόπηση στην Ουαλία και να ξέρουν οι Ουαλοί αν θέλουν να τους διοικεί το Westminster ή οι Βρυξέλλες. Ευχαριστώ κύριε Μπάφτον. Ο κύριος Γκολνής δεν είναι εδώ όμως, οπότε περνάμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Πίπερ για δύο λεπτά. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, τις ευρωπαϊκές περιφέρειες μια στιγμή ας τις φανταστούμε χωρίς την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική συνοχής. Πολλές πόλεις και περιφέρειες της Υπέδρου θα έχαναν υποστη... δυνατότητε για τις ε, διατωτικές αλλαγέ. Θα αφήναμε και θα εγκαταλείπαμε τις διαμεθοριακές περιοχέ, τι συνοριακέ περιοχέ. Η κοινωνική πολιτική δεν θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να έχει κονδύλια από την ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση ο μεσαίος τομέας ε, δεν θα ήταν δυνατό ε, να αντιμετωπίσει προβλήματα Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη χωρίς περιφερειακή πολιτική θα σήμαινε ότι η κοινότητα θα έχανε το πρόσωπό της, το χαρακτήρα της ε, στις περιφέρειες. Γι' αυτό είναι ανησυχητικά τα μηνύματα από την Επιτροπή ότι δεν θα, ήταν, ε, δεν θα υπήρχε η ανανέωση των ε, μέτρων συνοχής για, την, για τις περιφέρειες. Τι θα σήμαινε αυτό θα σήμαινε να χάσουμε τελείως ε, τη διασύνδεση και τη συνήφανση των ε, περιφερειών αυτών με την Ευρώπη. Θα γυρίζαμε στην εποχή της επανεθνικοποίησης. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τέτοια πορεία της ε, περιφερειακής πολιτικής δεν θα την υποστηρίξει με κανένα τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ε, δεν δεχόμαστε μεταρρυθμίσεις και δεν θα εξετάζαμε τέτοιες δυνατότητες. Με, τη, με τις αλλαγές και τις δημογραφικές αλλαγές ε, πρέπει να εντάξουμε τις, προσπάθειε προσπάθειές μας συγκεκριμένες αλλαγέ. αλλαγές θα πρέπει με μετρήσιμα μέτρα να, να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν με προσαρμογές. Περισσότερη χρηματοδότηση συν, περιφερειακά, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε προτάσεις από την Επιτροπή για την πολιτική που θα ακολουθηθεί. Αυτά τα μέτρα θα τα υποστηρίξουμε. Είμαστε αντίθετοι για την και τον κατακαιρματισμό και τη διάλυση της ε, περιφερειακής πολιτικής. Όχι στην επανεθνικοποίηση. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίπερ. Για 1,5 λεπτό θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Σταυρακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που πήραν το λόγο μέχρι τώρα και θα ήθελα να επισημάνω από την πλευρά μου και εγώ ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια πολιτική συνοχή μετά το 2013 που πρώτον θα κάνει διακρίσει μεταξύ των περιφερειών τη ευρωπαϊκή ένωση με προτάσει όπω κατάργηση του στόχου δύο ενδεκονιστικότητα δεύτερον θα περιέχει επανεθνικοποίηση πολιτικών και τρίτον θα αποκλείει του φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση από τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των κοινοτικών προγραμμάτων. αντίθετα οραματιζόμαστε μια πολιτική συνοχή για μετά το 2013 περίοδο που θα συνεχίζει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και θα εφαρμόζεται σε όλε τι περιφέρειες τη ευρωπαϊκή ένωση θα συνεχίζει να έχει ικανά χρηματοδοτικά μέσα για την εκπλήρωση του στόχου τη και θα έχει απλοποιημένου κανόνε εφαρμογή για να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία με προβλημάτισε το περιεχόμενο του εγγράφου για τη στρατηγική του 2020 γιατί δεν υπάρχει αναφορά στην πολιτική συνοχή ενώ είναι το κατεξοχήν κατάλληλο εργαλείο για την εκπλήρωση των στόχων τη Λισαβόνα και ήδη μεγάλο κομμάτι τη πολιτική συνοχή υπηρετεί αυτού του στόχου και έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία τη. Επίση, σημαντική απόδειξη για τη σημασία τη είναι ότι η πολιτική συνοχή απετέλεσε την αιχμή του δόρατο του σχεδίου ανάκαμψη τη ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια πολιτική ανάπτυξη μια πολιτική αλληλεγγύη μια πολιτική για κάθε ευρωπαίο πολίτη σε όποια περιφέρεια τη ευρωπαϊκή ένωση και να ζει. δυστυχώ όμω κάποιοι στην ευρωπαϊκή επιτροπή το ξεχνούν ή δείχνουν να το αγνοούν επεξεργαζόμενοι προτάσει που αλλάζουν τι αρχέ και τη μορφή τη πολιτική συνοχή. να είστε σίγουρο κύριε πρόεδρε όμω ότι εμεί θα του το υπενθυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία. σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τώρα θα λάβει το λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριος Τόιρερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ε, περιφερειακή πολιτική είναι μια πολιτική η οποία προβάλλει την Ευρώπη στις πόλεις, στις κοινότητες και στις περιοχές, ε, περιφέρειες υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συνεργάζονται και γι' αυτό η ολοκληρωμένη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρηθεί. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελλοντική Πολιτική συνοχής να ε, ασχοληθεί περισσότερο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εμπλέξει τις μικρές κοινότητες και τους δήμους ε, ή στην πολιτική συνοχής. Θα χρειαστούμε και στο μέλλον ε, επενδύσεις ή τις υποδομές, αλλά ιδίω καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο μέλλον θα πρέπει επίσης να προωθηθούν οι θέσεις εργασίας και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια τέτοια δομή της ε, πολιτικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Τόρερ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Ο κύριος Αλφόνση, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με ακούτε καλά, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ε, ομάδα των Πρασίνων η πολιτική αυτή είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Πρόκειται για την αλληλεγγύη. Η Ευρώπη ενισχύεται κάθε φορά που εκφράζεται η αλληλεγγύη και γι' αυτό είναι το θέμα αυτό βασικό για μας. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε τις εξής αρχές. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει πέραν της εδαφικής προτεραιότητας μια δημοσιονομική προτεραιότητα. Η βάση της ε, της ε, αναπτύξεως της περιφέρειας ε, είναι περιφερειακή άρα δεν μπορεί να επανενταχθεί σε εθνικό επίπεδο. Επίσης δεν θα πρέπει βασιστεί κανείς σε μεμονωμένα στοιχεία μιας περιφέρειας αλλά σε ένα σύνολο. λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πολιτική βέβαια διαφοροποιημένοι σύμφωνα με το επίπεδο πλούτου τους αλλά κάθε φορά που υπάρχει πολιτική συνοχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα θέματα. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Έρνστ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση έχει θεμελιώδη σημασία για τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση είναι η αγορά ή κοινωνική πολιτική θα πριτανέσουν. Οι προβληματισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής είναι απαράδεκτοι. Πρέπει να ενισχυθούν τα διαθροτικά ταμεία και όχι να συρρυκνωθούν. Και η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει λιγότερα, αλλά περισσότερα για την υπέρβαση, την αντιμετώπιση των περιφερειακών διαφορών. Το λέω κάθετα και απερίφραστα. Η επανεθνικοποίηση ακόμα και μέρους ή τμήματων της περιφερειακής πολιτικής θα είχε πάρα πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ε, για τη Γερμανία, για το ανατολικό της τμήμα και για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαφορές μεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξηθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λάβουμε υπόψη κοινωνικές, οικονομικές προϋποθέσεις ε, και όρους ε, για εκείνες τις περιφέρειες που έχουν το 50% ως τιμή κατοφλίου. Μία απότομη διακοπή αυτό, της, ε, των μέτρων στήριξης για αυτές τις περιφέρειες θα ήταν κάτι το πάρα πολύ αρνητικό. Επίσης η ενίσχυση των συγκεκριμένων ε, πόλεων και αστικών κέντρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση η υποστήριξη αυτή είναι πολύ σημαντική. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλο δυναμικό για την οικονομία και για τον οικονομικό τομέα. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει πλήξει η οικονομική κρίση αυτό το τομέα και ε, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει πάρα πολλά να επενδύσουμε, πάρα πολλά να κάνουμε και έχω ιδιαίτερες ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το κάνει και γι' αυτό έχει αποτύχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ένς. Για δύο λεπτά θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Όβερμαϊρ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εν τω μεταξύ θα και πληροφορηθεί υποθέτω ότι στην ε, Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το έγγραφο, το μυστικό κρυφό έγγραφο το οποίο κυκλοφορεί είναι διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το 2013 έως το 2020 μια αλλαγή πορείας κατά 180 μοίρες, μια απόλυτη ανατροπή των δεδομένων και μάλιστα το νέο σχέδιο προβλέπει τεράστια συρρήκνωση των μέτρων για την αρχή της επικουρικότητας και την ε, multi-governance και πράγμα το οποίο βρίσκεται σε αντίθεση με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Ιδιαίτερα σε σχέση με την αύξηση του στόχου 2, ανταγωνιστικότητα πολιτική ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τέτοιε περιφέρειες και περιοχές στόχου 2 στις ε, χώρες μέλη. Αυτό θα αφορούσε ιδιαίτερα και με αρνητικό τρόπο θα έπλητε τις περιφέρειες. Εδώ, σε σχέση με τα νέα κράτη-μέλη ή και με τα μελλοντικά λέει κράτη-μέλη, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που χρειάζονται νέα μέτρα, νέα κονδύλια και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ανακάμψει η οικονομία. Με αυτές τις προτάσεις βλέπουμε ότι ήδη μια ένταξη της ε, Τουρκίας ε, και η προοπτική αυτή και οι ανάγκες ε, που υπάρχουν οικονομικά, τεράστια κονδύλια τα οποία χρειάζονται θα πρέπει να διασφαλιστούν με αυτούς τους ελιγμούς. Το λέω όμως κάθετα ότι η περιφερειακή πολιτική εξαρτάται από την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να διατίθενται τα κονδύλια με αποτελεσματικό και λογικό τρόπο. Και αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα αντιμετωπίσουμε σωστά την οικονομική κρίση. Και δεν μπόρεσα να πιστώ από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, αναμένω συγκεκριμένη τοποθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Γκρέκ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μας ε, στηρίζει την πολιτική αυτή που θα επιτρέψει την ε, σύγκληση των ευρωπαϊκών περιοχών. Πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική πρέπει να ενισχυθεί και από κοινού το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή πρέπει να διαγράψουμε την πολιτική αυτή. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και τον προϋπολογισμό μετά το 2013 που θα πρέπει να εμπλέξει όλους τους ενδιαφερόμενους την περιφέρεια, τις περιφέρειες, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να αποδυναμωθούν τα τοπικά σκέλη που δίνουν νόημα σε αυτή την πολιτική. Από πλευράς δημοσιονομικής σήμερα έχουμε μια μεγάλη ασάφεια όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής διότι ε, το τέλος του τωρινού πλαισίου είναι άγνωστο και αβέβαιο και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι χρειαζόμαστε μία συνεχή χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε μία επανεθνικοποίηση αυτών των ε, πολιτικών που θα ε, εξουδετέρωνε τη διάσταση που χρειαζόμαστε της πολιτικής αυτής. Πρέπει να είμαστε θετικοί, να προετοιμάσουμε μία λευκή βιβλό για την ε, εδαφική συνοχή. Δεν θέλουμε να υπάρχει τεχνητή ισότητα αλλά ουσιαστική και να τονίζονται οι, οι διαφορές των ε, περιοχών. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μόνο τις πιο φτωχές ε, περιοχές αλλά όλες και ιδίω ε, τις υπερπόντιες. Θα πρέπει να μιλάμε με σταθερούς και συγκεκριμένους ομολόγους κατά τρόπον ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να κατανέμονται δίκαια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Γκρέκ. Τώρα, για ένα λεπτό, ο κύριος Κορτές, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι σε σχέση με τις κοινωνικές αυτές εκφράσεις στην Κοπεχάγη και να χαιρετήσουμε για το μέλλον της ε, ε, πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια ισχυρή ε, πολιτική συνοχή και να είμαστε κατά της επανεθνικοποίηση για την ανάπτυξη των κρατών μερών, αλλά επίσης και όσον αφορά την στρατηγική για τη σταθερότητα, την χρηματοοικονομική και τον ευδιάκριτο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ο ρόλος τον οποίο θα πρέπει να αναπτύξουν οι περιφέρειες μέσα στην περιφερειακή, πολιτική συνοχή. Είναι σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη τη ε, ε, πολιτική συνοχή. Επίση, όσον αφορά την μεταβατική περίοδο που θα διασφαλίζει την ε, περίοδο αυτή για τα κράτη Κίνα, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε σχέση με του στόχου συνοχή και του στόχου των διαθροτικών ταμείων, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιομορφίε των ιδιαίτερων περιοχών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Κορτέ. Για ένα λεπτό η κυρία Φιγκερέδο παρακαλώ. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις ε, τις δημοσιονομικές του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαθροτική πολιτική και την πολιτική συνοχή, Σε μια κατάσταση κρίσης και μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων, η πολιτική, η διαρθρωτική και η συνοχή είναι θεμελιώδου σημασία ε, για την ε, κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερα με συγκεκριμένους στόχους σε αυτόν τον τομέα. Και όχι να προσπαθούμε να επανεθνικοποιήσουμε το κόστος της κοινωνικής πολιτική, είτε στην γεωργία, είτε ασκείται στην Αλία, δίνοντας αρνητικές επιπτώσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Υπάρχουν όμως αρκετές ενδείξεις ότι θέλουν ακόμα περισσότερο να ανατρέψουν τις αρχές ε, αυτές. Όσον αφορά την χρηματοδότηση ε, δράσεων που δεν έχουν καμιά σχέση με τους στόχους συνοχής, ιδιαίτερα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000, μέχρι το 2020 και όσον αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών κλιματικών αλλαγών όσον αφορά κριτήρια διαχείρισης για αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό έχει κάθε νόημα να γίνει αυτή η συζήτηση για την πολιτική συνοχή μετά το 2013. Αναμένουμε σαφείς απαντήσεις για μια πραγματική πολιτική κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για δύο λεπτά ο κύριος Τεσέιρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Είναι κατεπήγον να γίνει αυτή η συζήτηση σε σχέση με τις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωση και το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την αηφορία και τη διαφάνεια. Για το πλαίσιο μετά το 2013 πρέπει με βάση την αλληλεγγύη και την περιφερειακή συνοχή να δράσουμε με ε, βάση αυτές τις θεμελιώδεις αξίες για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Θέλω να συμμεριστώ μαζί σας κάποιες ιδέες που θεωρώ ότι πάντα πρέπει να μας προβληματίζουν όταν οικοδομούμε την πολιτική συνοχή. Η συνοχή που αναφέρεται επανειλημμένα, κάποιες πτυχές θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η ελαστικότητα, η απλούστευση, η αποτελεσματικότητα και η επίτευξη των στόχων που έχουν προβλεφθεί. Υπάρχουν θέματα όμως τα οποία δημιουργούν κάποιες ανησυχίες, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπερπεριφερειακών περιοχών περιοχών, των πιο απομακρυσμένων δηλαδή περιοχών. Ιδιαίτερα όσον αφορά την προσέγγιση αυτών των περιοχών πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ δράσει όπω ε, ο τομέα πρόσθετη ε, αξία. Πρέπει εδώ να δούμε ότι δεν πρέπει να, να αμφισβητηθεί, να υπονομευθεί ο στόχο 2. Ε, πρέπει να δούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε αντιπαραγωγικοί σε υπεραπομακρυσμένε περιοχέ. Δεύτερο, θεωρώ ότι η διατήρηση τη αρχή τη προσέγγιση στην πολιτική πολιτική αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε υποπεριφερειακό πρίσμα τα κονδύλια για την διαθροτική ανάπτυξη και όχι υποκεντρικό πρίσμα. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω το άρθρο το 349 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Προβλέπει ειδική αντιμετώπιση των απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαθροτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την μειονεκτική τους ε, κατάσταση όσον αφορά την απομάκρυνση, και την οικονομική ε, συγκυρία. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, εξειδικευμένη υποστήριξη που θα διαθέσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τεσέρα. Για ένα λεπτό θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Ολέχνιτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή σήμερα βοηθάει τα νέα κράτη-μέλη να αναπτύξουν υποδομές, ε, δρόμους, υδροδρόμους, Χάρη σε αυτή την πολιτική θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στο μέλλον. Επενδύσεις για το περιβάλλον επίσης που είναι πολύ σημαντικές. Στην αξιολόγηση της μέχρι τώρα πολιτικής θα έπρεπε κανείς να θέσει το ερώτημα τι θα γίνει μετά το 2013. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ε, δηλώσει σαφώς ότι δεν συμφωνούμε με την επανεθνικοποίηση θυμάτων της πολιτικής αυτής μετά το 2013. Ε, μέχρι στιγμής, πέραν των παραδοσιακών δράσεων και των παραδοσιακών μηχανισμών, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι επιστήμε, η καινοτομία, ποιοτικέ θέσει εργασία και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στις περιοχές της υπαίθρου. Είναι σημαντικό η πολιτική συνοχής να εφαρμοστεί ε, με βάση τις περιφέρειες και τις μακροπεριφέρειες. Σας ευχαριστούμε κύριε Λέχνιτσα. Ο κύριος Ντόιτς τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα πολύ γρήγορα. Στην δικαιοσύνη, στα μυστικά και τη σημασία της Ανάπτυξη της υπαίθρους. 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους ε, του Βερολίνου και από όταν ε, στην ε, τη Μισοάρα στη Ρουμανία ακούστηκε η φωνή του Λάσλο δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι τώρα δεν υπάρχουν πλέον παλιές και νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, θα μπορέσουμε να ε, ε, ε, υπάρξει μια κίνηση συμβολική αλλά επιπλέον και ουσιαστική στην, πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν τα κράτη-μέλη είναι ίσα δεν μπορούμε να φανταστούμε μια πολιτική διαφορετική και δεν θα πρέπει να είναι χαμένη οι χώρες που προσχώρησαν το 2004 και 2007. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια μεθαρρύθμιση. Είναι δηλαδή απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει δηλώσεις χωρίς ουσία ή να σιωπά. Σαν Ευρωβουλευτές και σαν μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαντάζομαι ότι και εγώ μπορώ να ζητήσω να έχω μία σαφή εικόνα. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο πολύ ουσιαστικό της αναπτύξεως και χρειάζεται πόρους για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η εξέλιξη αυτή. Είναι επίσης πολύ βασικό να μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε ε, ε, από το 2013 στην περιτροφή συνοχή στην ε, την πολιτική αναπτύξεως. Ο κύριος Άλβες, η πολιτική συνοχή είναι το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις για ευημερία όπου και αν ζουν. Επίσης η δημιουργία της, ε, ε, του αισθήματο του ότι ανήκουν στην Ευρώπη και είναι η καλύτερη δυνατότητα για να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη. Δεν μπορώ να κρύψω κύριε Επίτροπε την ανησυχία μου για αυτό το περιβόητο non-paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτάσεις του. Δεν δεχόμαστε την επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής η αποτελεσματικότητα έτσι θα εξαρτάται από, την, ε, από τον πλούτο του κάθε κράτους. Ελπίζω ότι θα εγκαταλείψετε αυτή την οδό από την Επιτροπή. Όπως ξέρετε το άρθρο 349 της Συνθήκης θέτει την ανάγκη της προσαρμογής ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών στις ανάγκες των απομακρυσμένων περιοχών. Ε, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και την χρήση του δυναμικού τους. Και έτσι λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε για τη μελλοντική στρατηγική και να υπάρξει η προσαρμογή αυτή αυτών των αρχών το 2010. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Άλβες. Και τώρα θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Κέλλη. Ε, thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοί μου, ανησυχώ και εγώ για κάποιες από τι τάσει που εμφανίζονται στο εσωτερικό έγγραφο και οι τομεί που μου προκαλούν τι μεγαλύτερε ανησυχίε είναι η πρόταση να επανακτικοποιηθεί, ε, να δοθούν μάλλον ε, άλλοι άλλες προτεραιότητες στους ε, διαφορούς στόχους σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Επίσης, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες στην έξυπνη οικονομία, όπως λέγεται, και αυτό θα πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη ένταση. Ε, στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι με, ανάμεσα στις περιφέρειες υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την φτώχεια. Και αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια που βασίζονται στο εθνικό ΑΕΠ είναι λανθασμένος τρόπος μέτρησης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη που σε ορισμένες περιφέρειες είναι πολύ πιο χαμηλή από ότι ο εθνικός μέσος όρος. Ε, πρέπει λοιπόν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες συνέργειας που υπάρχουν ε, ανάμεσα στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην πολιτική συνοχή. Και η περιοχή ανάπτυξης της υπαίθρου είναι ένας σημαντικός παράγοντας και δεν θα πρέπει να συρρυκνωθεί σε οποιασδήποτε μελλοντικέ ε, προτάσεις, διότι η ανάπτυξη της υπαίθρου και τα οικογενειακά αγροκτήματα είναι ζωτικής σημασία για την ε, ε, επιβίωση της κοινωνίας αυτής. Ξέρω ότι πρόσφατα έχουν πραγματοποιηθεί βήματα ε, βελτίωσης, αλλά πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πηγαίνουν πραγματικά στους πραγματικούς αποδέκτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Λοιπόν, προσέξτε κυρίες και κύριοι τώρα. Τώρα θα περάσουμε στον γύρο των ετοιμάτων για παρέμβαση από πλευράς των Ευρωβουλευτών Catch the Eye. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν τον λόγο. Γι' αυτό να μην ζητήσετε περισσότεροι να παρέμβετε, διότι έχει κορεστεί ο αριθμό ήδη. Για ένα λεπτό θα λάβει τον λόγο η κυρία Λουκασεύσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι εκπροσωπώ την περιφέρεια του Πορτ Καρπάτσε στην Νότια Πολωνία. Είναι μια ε, περιφέρεια με πολύ δυναμικό κόσμο και επιχειρήσεις όπου υπάρχουν ε, νέα επιχειρηματικά κέντρα όπως ε, η λεγόμενη ε, κοιλάδα της ε, αεροπορίας. Η υπόλοιπη όμως περιφέρεια είναι σχετικά φτωχή. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε λοιπόν αυτή την φτώχεια μέσω μιας σειράς προγραμμάτων. Δεν χρειαζόμαστε όπλα, δεν χρειαζόμαστε ελεημοσύνη, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες λύσεις που θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Θέλουμε οποιασδήποτε ε, αλλαγέ στι ε, προτεραιότητε όσον αφορά τη χρηματοδότηση να γίνουν με ομαλό και σταδιακό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να είναι οι περιφέρειε αυτέ που θα εφαρμόζουν την πολιτική συνοχή. Αυτό δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Επίση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα μήνυμα προ του πολίτε τη Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Φερχέγγεν, παρακαλώ. Η περιφερειακή διαρθρωτική υποστήριξη είναι ένα ουσιαστικό μέσο για την περιφερειακή συνοχή. Και στο παρελθόν ως κινητήρας για την διαθροτική και οικονομική ανάπτυξη σε πολλές περιφερειές χρησιμοποιήθηκε υπέρ των ανθρώπων. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των προσαρμογών και των αναγκαίων δράσεων και για τις κοινότητες εδώ, για την Ευρώπη των πολιτών επιτόπου αυτό μπορεί να το δει κανείς χειρόπιαστα. Χρειαζόμαστε όμως μια πιο σαφή και πιο διαφανή δομή στα ταμεία συνοχής, στα κονδύλια συνοχής, ώστε τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται με αηφορία και αποτελεσματικότητα για την ε, προσαρμογή και την ε, ανάπτυξη την οικονομική που είναι κύριοι στόχοι θα πρέπει αυτά τα μέσα όχι να τα αποδυναμώσουμε στο μέλλον αλλά να τα ενισχύσουμε. Η πολιτική συνοχή στην Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να παραμείνουμε στα συστήματα σορευτικότητα ή προσθετικότητα. Δεν θέλουμε πανεθνικοποίηση για την ενίσχυση. Γι' αυτό παρακαλούμε τα κριτήρια το, για το, ε, μετά μετά το 2013 να ληφθούν αυτά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Φόερ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ουαλία είναι ίσως η πιο, ε, το πιο καλό παράδειγμα περιφέρειας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό γιατί ε, όλοι υποφελούνται από την ε, Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, πρώην στόχο 1, τώρα ε, από το, τα τη χρηματοδότηση για την σύγκληση. Ε, θα πρέπει η Κομισιόν να λάβει υπόψη τι συνέπειε θα έχει ο απονομισμό των στόχων για περιφέρειε όπω η Ουαλία. Ε, να σκεφτούμε τι οικονομικέ ε, και κοινωνικέ ε, συνέπειε για τι περιφέρειε αυτέ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία όλοι οι Ευρωβουλευτέ να παροτρύνουν την Κομισιόν να υποβάλει προτάσει που θα είναι αποδεκτέ ε, για μα. Και με αυτό εννοώ προτάσει οι οποίε θα επιτρέπουν κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη που έχει και πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια να ε, έχει πρόσβαση στα διορθωτικά ταμεία. Και αυτές που είναι έξω από την σύγκληση ε, του 2013 ε, να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και για αυτές. Σας ευχαριστούμε κύριε Βόν. Κύριε Γκόλνης φτάσατε τώρα επιτέλους έτσι. Λοιπόν, θα έχετε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις επεμβάσεις των συναδέλφων. Νομίζω ότι καταλήγουμε ουσιαστικά σε δύο συμπεράσματα. Καταρχήν την μυστικότητα ε, αυτού του μη εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία της εξηγής της Επιτροπής και δεύτερον το περίεργο γεγονός ότι θα αναπροσδιοριστεί η πολιτική εδαφική συνοχή γύρω από νέου άξονες οι οποίοι φαίνονται να έχουν ελάχιστη σχέση με αυτή τη συνοχή. Εδώ αναφέρομαι στην εξωτερική πολιτική που ξέρουμε ότι είναι προτεραιότητα για τον ύπατο εκπρόσωπο αλλά πολύ λιγότερο σε αυτό το τομέα. Για την κοινή γεωργική πολιτική ήδη έχει θυσιαστεί στους νόμους της αγοράς και πιστεύουμε ως εκ τούτου ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει σαφώς ποιοι είναι τώρα οι στόχοι της και για την ε, θέρμανση της, ε, ε, του κλίματος που δεν εξαρτάται από την πολιτική συνοχή. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Παλώνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις ανησυχίες πολλών συναδέλφων. Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση με ρυθμούς ανάπτυξης μόλις θετικούς για το 2010 ε, θα ε, έχει λήξει ε, και θα φτάσουμε σε επίπεδα απασχόλησης όπως πριν από την κρίση. Ε, αναφέρομαι στο 2010. Και γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική επενδύσεων και είναι πολύ σημαντικό ο στόχος 2 να διατηρηθεί ή κάτι παρόμοιο με το στόχο 2 διότι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο ε, που βοηθάει τις ε, περιφέρειές μας να ξεπεράσουν την κρίση. Η διατήρηση του στόχου 2 ε, είναι κάτι που αφορά και την Ιταλία και πολλές άλλες χώρες. Είναι μια ουσιαστική απέτηση. Η εξέλιξη των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση για να φτάσουν τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες η εγκατάλειψη του στόχου 2 θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τι περιφέρειες τη Ιταλία, τη Ευρώπη και τη Μεσογείου και άλλων χωρών. Σα ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ κύριε Παλώνε. Τώρα για ένα λεπτό Ρέγνερ παρακαλώ. Η κυρία Ρέγνερ. Η κυρία Ρέγνερ παρακαλώ. Πολλοί μιλούν για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, αλλά στην Ευρώπη αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην πολιτική συνοχή. Γι' αυτό θα ζητούσα μία ανεξάρτητη πολιτική ε, και ε, να ενισχυθεί το κοινωνικό ταμείο, το οποίο να είναι πιο ισχυρό και να υπάρξει αποθήκευση πόρων για την μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο, κατά τρόπον ώστε στην πολιτική αυτή να μπορέσουν να διατεθούν επαρκή σπόροι σε περιοχές οι οποίες χρειάζεται να καλύψουν τα κενά και που δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής ε, ε, υπόψη από τις πολιτικές. Θα πρέπει συγχρόνως το Ταμείο αυτό να καλύψει τα θέματα ανεργίας, ε, εγκατάλειψη των, των σχολείων από τους μαθητές και βελτίωση των συνθηκών. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρέγνερ. Για ένα λεπτό κυρία Κράτσα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θεωρώ πολύ σημαντική την απόφαση της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής για αυτή τη συζήτηση σήμερα η οποία αποδεικνύεται και πολύ ενδιαφέρουσα αφού τέθηκαν τόσα ζητήματα διαστάσεις ε, ε, πολύ σημαντικές που αφορούν όχι μόνο μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής μετά το 2013 αλλά και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συζήτηση αυτή, ο προβληματισμός αυτός διατυπώνεται σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια μεριά έχουμε ένα βήμα θετικό προ την ολοκλήρωσή τη με τη συνθήκη τη λισαβόνα από την άλλη πλευρά βιώνουμε ακόμη τι συνέπειε μια πρωτοφανού χρηματοπιστωτική κρίση διεθνού που όλοι αντιληφθήκαμε πόσο σημασία έχει η αλληλεγγύη τη ευρωπαϊκή ένωση για την υποστήριξη της εσωτερική αγορά και τη σύγκληση. θα ήθελα ε, και εγώ να ρωτήσω ε, την ευρωπαϊκή επιτροπή να μας ε, κάνει μια σαφή δήλωση για δύο θέματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. συμμερίζομαι με τον συναδέλφον τον προβληματισμό. αν υπάρχει στους σχεδιασμούς σας για καινοτόμες προτάσεις που θα τις δεχτούμε ευχαρίστως με αν υπάρχει η διάθεση επανεθνικοποίησης της πολιτικής της συνοχής και δεύτερον το μέλλον του στόχου 2 γιατί είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται την ανταγωνιστικότητα όχι μόνο ορισμένων περιοχών αλλά τελικά του συνόλου της ευρωπαϊκής αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κράτσα. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Κάλμαχ παρακαλώ. Κυρία Κάλενμπαχ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έργο μας εδώ ως Ευρωκοινοβούλιο και έργο της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες πλαισίου ώστε οι πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη στις περιφέρειες όπου ζουν να έχουν την ανώτατη ε, αναμενόμενη ποιότητα ζωής. Οι προϋποθέσεις όμως γι' αυτό στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικές και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής με προβληματισμούς που ακούσαμε να παρουσιάζονται που θα σημαίνουν ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη πορεία. Όχι, δεν χρειαζόμαστε επανεθνικοποίηση, δεν χρειαζόμαστε ανατροπή πορείας, χρειαζόμαστε μέσα στήριξης για όλες τις περιφέρειες, για όλους ε, που έχουν συμμετάσχει και έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικά. Δεν μπορούμε το κεκτημένο να το υπονομεύσουμε. Χρειαζόμαστε ένα διαφανέ σύστημα χρηματοδότησης που θα διευκολύνει την πρόσβαση, από την άλλη όμως πλευρά θα διασφαλίζει ότι τα χρήματα, τα κονδύλια κονδύλια θα, ε, θα διανέμονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάντενμπαχ. Τώρα στη συνέχεια για ένα λεπτό ο κύριος Ματούλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ε, ακριβώς γιατί λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση. Οι αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών ε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι περιφέρειες αυτές χρειάζονται μια συνέχιση της πολιτικής συνοχής. Η μείωση των ε, διαφορών μεταξύ των διαφόρων περιφερειών πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορα, δεν πρέπει να επιβραδυνθεί. Βεβαίω, η συμμετοχή των επιπέδων διακυβέρνηση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να ενισχυθεί. Οι περιφέρειε όμω δεν πρέπει να ε, αισθανθούν ότι σιγά σιγά εγκαταλείπονται από την Ευρώπη. Πολλέ χώρε βασίζουν τι αναξιοπτικέ του προσπάθειε και τι εθνικέ του πολιτικέ ε, και μάλλον στα πλαίσια πλαίσια αυτά λαμβάνουν υπόψη τους και συνυπολογίζουν την πολιτική συνοχής. Ε, υπάρχει λοιπόν η ελπίδα ότι θα συνεχιστεί η πολιτική συνοχή μετά το 2013 σε συνδυασμό και με το κοινωνικό και με το περιφερειακό ταμείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ματούλα. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Παπαδοπούλου, Παπαδοπούλου Πρόεδρε, θα συμφωνήσω πως η περιφερειακή πολιτική είναι κινητήριος μοχλός για καλύτερη κοινοτική συνοχή και αλληλεγγύη. Η παρούσα διεθνής οικονομική κρίση έχει τρίξει τα δόντια. Δημιούργησε αρκετές ανισότητες και πιέσεις, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες αύξησε την ανεργία τι ανισότητε την κοινωνική αναστάτωση σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό. η παρούσα διεθνή οικονομική κρίση συνιστά όμω και μια πρόκληση υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση τη κοινωνική αλληλεγγύη για μια σωστή και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική συνοχή που να θέτει ψηλά προτεραιότητε να διασφαλίζει σωστέ υποδομέ και στενότερη διασυνοριακή συνεργασία με ανταλλαγή καλών πρακτικών. λέμε όχι στι διακρίσει όχι στην επανεθνοποίηση επανεθνικοποίηση όχι στη γραφειοκρατία όχι στην αδιαφάνεια όχι στη μυστική διάθεση κονδυλίων και στην κατάργηση του στόχου 2 που θα πλήξει τη νότια ευρώπη και τη μεσόγειο. λέμε ναι στην ακριβοδίκαιη κατανομή των κοινοτικών πόρων στη συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις σωστές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση δράσεων που θα συνάδουν με στόχους της για το 2020 Λέμε ναι και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε στην ειδική αντιμετώπιση απομακρυσμένων περιοχών, ιδίω στην Νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Λούχαν παρακάτω Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αύξηση της διακυβέρνησης σε πολλά επίπεδα δημιούργησε διάφορες πλατφόρμες και οι τοπικές αρχές πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγάλες διαφορές ε, όσον αφορά τις πολιτικές ε, τις οποίες δεν ελέγχουν και τις οποίες δεν επηρεάζουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επηρεάσει κανείς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ε, προγραμμάτων τα οποία εφαρμόζονται συγχρόνως σε διάφορα επίπεδα. Θα ήθελα να ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βοηθήσει τις τοπικές αρχές και να εφαρμόσει μία συνεκτική στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες οι οποίες μπορεί να έχουν αλλάξει ή <clears throat> να έχουν επηρεαστεί από εξωτερικές αιτίες. Δηλαδή ε, τι μέτρα θα χρησιμοποιηθούν για την ε, εφαρμογή από τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ κύριε Λούχαν. Κλείνουμε τον γύρο των ε, συζητήσεων αυτό με τον κύριο Σικέρσκι για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η πολιτική συνοχή αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής ανάπτυξης της Ένωσης. Η πολιτική αυτή ενισχύει περαιτέρω τις τοπικές αρχές και τις περιφέρειες. Στην αξιολόγηση αυτή, ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε δύο ακραία ε, ενδεχόμενα. Να περιορίσουμε πολύ την πολιτική συνοχή ή να την επεκτείνουμε ιδιαίτερα πρέπει να έχει μια ισορροπημένη προσέγγιση πολιτική συνοχής και για τις αστικές περιοχές και για την Ήπεθρο. Μετά την διεύρυνση, η Ένωση έχει ακόμα μεγαλύτερες εσωτερικές ανισότητες που πρέπει να επιτρέψουν να υπάρχει ε, ε, ίδια αντιμετώπιση όλων και για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση πρέπει να λάβουμε υπόψη τις οικονομικές τάσεις και τις αλλαγές του κλίματος. Κάτι που είναι βέβαιο ωστόσο είναι ότι χρειάζεται να συνεχιστεί η πολιτική συνοχή και να προσαρμοστεί στι υφιστάμενε προκλήσει. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε χρόνο και πρέπει να είμαστε και ευέλικτοι και καλοσυνάτοι λόγω της εποχής. Δίνω το λόγο στην κυρία Τικάου για ένα λεπτό. colegul meu faptul că atunci când vorbim de orașe inteligente este important să όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, όταν μιλούμε για έξυπνες πόλεις πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Το 90% των κτηρίων που θα υπάρχουν το 2020 υπάρχουν ήδη και τώρα, που σημαίνει ότι η πολιτική της Επιτροπής θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη ποσόστοση των πόρων περιφερειακής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη για χρήση ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και των σπιτιών. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να επενδύουμε περισσότερο στην, ε, στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Ήμουν καλός με την κυρία Τικάου. Θα είμαι και με τον κύριο Παπα-Νικολάου. Θέλετε ένα λεπτό κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοί μου έχουν καλύψει τα βασικά θέματα της σημερινής μας συζήτησης. Θα ήθελα να δώσω έμφαση σε δύο μόνο θέματα. Το πρώτο, δεν είναι δυνατόν σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες για να αξιοποιηθούν οι πολιτικές μας και τα προγράμματά μας για τη συνοχή και τελικά για λειτουργικούς λόγους και κυρίως γραφειοκρατικούς αυτό να μην γίνεται εφικτό. άρα λοιπόν όσο απλουστεύουμε τις διαδικασίες μας και τις πολιτικές μας τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε αυτό που επιδιώκουμε στη συνοχή της ευρώπης. το δεύτερον είπαμε ότι βαδίζουμε ούτως ή άλλως προ την έξοδο από την οικονομική κρίση που ταλανίζει όλη αυτή την περίοδο την ευρώπη και όλο τον κόσμο. αν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι είναι δεδομένο ότι πρέπει να ενισχύσουμε εκείνε τι περιοχέ που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και κυρίω αν μου επιτρέπετε και σε αυτό θα ήθελα μια απάντηση από την επιτροπή εκείνε τι κοινωνικέ ομάδε που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ενδυνάμωση και αναφέρομαι κυρίω στου νέου αυτή είναι η βασική μας θέση και ειδικά της πολιτικής μας ομάδα σε σχέση με την κοινωνική οικονομία της αγοράς και μόνο έτσι μπορούμε να ατενίζουμε με σιγουριά το μέλλον. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπα-Νικολάου. Το λόγο έχει για την Επιτροπή ο Επίτροπος κύριο Σαμέτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση της ε, Ατζέντα 2020, μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα ανταποκριθεί σε πολλές ε, προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η πολιτική συνοχής, που θα είναι και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ως εκ τούτου ανησυχίε ότι η πολιτική συνοχή ε, θα αποχωριστεί από την συνολική εφαρμογή και υλοποίηση της στρατηγικής αυτής είναι αβάσιμες. Δεύτερον, σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη φάση, πολλές ερωτήσεις και πολλά ζητήματα, επί παραδείγματι γεωγραφική κάλυψη, οι περιοχές στόχου 2, κατάλληλη βάση, μεταβατικές ε, διευθετήσει με μονομένες ε, περιφέρειες ή ομάδες περιφερειών κτλ. Τέτοια θέματα τα οποία ε, τέθηκαν και από τους αξιότιμους βουλευτές παραδέχομαι ότι δεν έχουν απαντηθεί σαφώς ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σε βάθος συζήτηση μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μεταξύ κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων και εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση αυτή θα οδηγήσει στην εκπόνηση της μακρόπνοης θέσης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010. Τους προσεχείς μήνες τα ζητήματα και τα προβλήματα που τέθηκαν εδώ θα τύχουν τη σωστή κατάλληλη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν τέλει, θα ήθελα να ευχαριστήσω του αξιότιμου βουλευτέ για τι ερωτήσει του, για τι υποδείξει του οι οποίες επιβεβαιώνουν τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως ενός εργαλείου ε, και μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης, αν θέλετε, ε, για την ανάπτυξη του δυναμικού των ε, περιφερειών και των κρατών μελών. Λαμβάνω υπόψη τα σχόλιά σας, τις υποδείξεις σας και θα τα διαβιβάσω όταν επιστρέψω στις Βρυξέλλες στους συναδέλφους μου από την ε, δική μου γενική δένση και στον ε, Επίτροπο που θα με διαδεχθεί στα καθήκοντά μου και ελπίζω ε, τους επόμενους μήνες να έχετε την πρόταση αυτή για την πολιτική Σας Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το σημείο της μετρησιάς διάταξης. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 11.30 οπότε και θα λάβει χώρα η ψηφοφορία.